Test um, dois, Test Test um, dois, test um, dois. test um, dois. Τεστ, unser corona With the Αναζήτησε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 να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα από την πρώτη ψηφοφορία και μετά να περάσουμε στη δεύτερη γύρω ψηφοφοριών. Τα αποτελέσματα λοιπόν σε ό,τι αφορά τις, ε, τα αιτήματα για διαδικασίες κατεπήγοντος. Δεν θα τα διαβάσετε τα αποτελέσματα, θα τα βρείτε στην οθόνη σας. Τώρα έχουμε για τον κανονισμό για την πρωτοποίηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Με διαδικασία κατεπήγοντος λοιπόν εγκρίθηκε η διαδικασία κατεπήγοντος. Αυτοί που ακούνε από έξω δεν βλέπουν την ε, οθόνη. 684 οι ψήφοι, 670 υπέρ, 13 κατά, μία αποχή. Τώρα έχουμε το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού αριθμός 1 στο 2020. Εγκρίθηκε επίσης. 684 ψήφοι συνολικέ, 658 υπέρ, 7 κατά, 19 αποχέ. Σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού εδαφμό υπαριθμό 2 του 2020, παροχή στήριξη έκρηξη ανάγκη στα κρατημέλη επίση εγκρίθηκε. 684 οι ψήφοι, συνολικά 678 υπέρ, 5 κατά, μία αποχή. Τώρα έχουμε την ε, κινητοποίηση του Μηχανισμού Ευελιξίας για το 2020, το έγγραφο 2020, κάθετος 2053. Επίσης εγκριθήκαν ε, οι διαβουλεύσεις για τη διαδικασία κατεπήγοντος. Τώρα περάσαμε στο δεύτερο α, μηχανισμό ευελιξίας. Θα ήθελα παρακαλώ το 2020-2053, λέει ο, ο πρόεδρος. Το 2020 κάθετος 2053 λεει ο ο το 2020 καθετος 2053 μηχανισμός ευελιξίας υπαριθμών 1. Δεν θέλω το δεύτερο, λέει ο πρόεδρος. Έχω μόνο τον αριθμό του εγγράφου. Το 2020 κάθετος 2053. Το υπαριθμό 2 είναι το 2020-2056. 684 λοιπόν οι ψήφοι. Συνολικά. 657 οι ψήφοι υπέρ, 8 κατά, 19 αποχές. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν τώρα το έγγραφο 2020 κάθετος 256. 684 συμμετείχαν, 664 υπέρ, 6 κατά, 14 αποχές. Έχουμε τώρα την ε, τοποίηση του περιθωρίου για προβλήτες ανάγκες. Εγκρίθηκε η διαδικασία κατεπήγοντος. Για τις απρόβλεπτες ανάγκες, παρακαλώ, υπάρχει το έγγραφο. όχι για το COVID-19. Μηχανισμός ευελιξίας υπαριθμών 2. Θέλουμε τώρα τις απρόβλεπτες ανάγκες, τις απρόβλεπτες δαπάνες κινητοποίηση στην περιφερεια για τις απροβλήτες ανάγκες. It is that unforeseen expenditures? Spielraums, yeah. Okay, also. Εδώ έχουμε λοιπόν 684 συναδέλφους που συμμετείχαν, 679 υπέρ, 4 κατά, αποχές 1. Εγκρίθηκε λοιπόν. Περνάμε λοιπόν στα ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διευθυντικών και Επιβεβαιτικών Ταμείων. Και τώρα τα βλέπουμε και στην οθόνη. 684 ψήφοι, 680 υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές και άρα εγκρίνεται το αίτημα για πηγών. Έχουμε θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19. 684 ψήφοι, 680 υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές και εδώ εγκρίνεται λοιπόν η διαδικασία κατεπήγοντος. Τώρα περνάμε στα ειδικά μέτρα για το μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της αλίας και της υδατοκαλλιέργειας. 684 ε, συμμετείχαν. 663 υπέρ, 615 κατά, 15 εποχές. Και εδώ λοιπόν εγκρίνεται η διαδικασία και κατεπήγον. Περνάμε στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 684 ψήφοι. 679 υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές και εδώ εγκρίνεται λοιπόν το αίτημα για κατεπήγουσα διαδικασία. Για όλε αυτέ τι κατεπήγουσε διαδικασίε έχουμε τώρα ε, προθεσμία 12 λεπτών μέχρι τις 2 για τις ε, τροπολογίες και σήμερα στις 3 15 ε, και 30, 3,5 θα έχουμε περιθώριο για τι διαχωριστέ ψηφοφορίε και θα ανακοινωθούν αύριο τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά για τα κοινά μέτρα για τις Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη πανδημία COVID-19 θα λάβει η χώρα στι 5. Και περνάμε τώρα στο δεύτερο γύρο ψηφοφοριών για τον κανονισμό για την τροποποίηση του πολιτού του δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και στο δεύτερο τμήμα των τροπολογιών για την συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών τη με την ίδια διαδικασία. Όπως σήμερα το πρωί, η δεύτερος γύρος ψηφοφορία μέχρι τι 4.30. Έχετε λοιπόν χρόνο μέχρι τι 4.30 για να ψηφίσετε. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στι 5 ε, και έτσι διακόπτεται η Σύνοδο.